λόγω, Σε γενικές γραμμές συζητάμε, έχουμε κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις. Τώρα, να σας πω που έχουμε διαφορετική άποψη σε μικρό βαθμό βέβαια. Ρωτάμε. Ε, Mr. Luca proposes some, ε, some figures. Γιατί. Ε, βάζει και κάποια αριθμητικά στοιχεία ο κύριος Λούκε. Και εδώ μιλάμε για τις μεταβλητές επί της ονομαστικής Τη ονομαστική αξία των στοιχείων ενεργητικών που μπαίνουν στο pool και εδώ έχουμε το 90, 80 και 60% ως ποσοστά και συντελεστέ. Και αυτές οι αξίες ε, πιστεύω που μπαίνουν στο πουλ λέει ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε αυτά τα ποσοστά. Εγώ ρωτώ, με ποιο τύπο υπολόγισε αυτά τα ποσοστά και γιατί έχουμε καταλήξει στο 90, 80, 60 και δεν έχουμε ας πούμε 85, 80, 75. Να σας πω πως έχουμε και μια-δύο ακόμα περιπτώσεις όπου και πάλι έχουμε αναφορά σε αριθμητικά στοιχεία, έχουμε τη στάθμιση ας πούμε για τις περιπτώσεις της επέκτασης χρονικής οριμότητας και πάλι έχουμε αυτά τα 5, 10, 15, 20 ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της επέκτασης της παράτασης, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι βασίστηκε για να καταλήξει αυτά τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Επιτάχυνση, τροπολογία 21. Επιτάχυνση πληρωμών σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας για τις πληρωμές οι οποίες έχουν, είναι εγγυημένε από αυτές τις καλυμμένες ομολογίες. Εδώ θέλουμε να το αφήσουμε ανοιχτό, να υπάρχει μια δυνατότητα ο επενδυτής να μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διάρκεια της επιτάχυνσης. Γιατί η τρέχουσα διατύπωση δεν δίνει καμία δυνατότητα για τον επενδυτή να επηρεάσει την ταχύτητα αποπληρωμή σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα. Και για την ομοιογένεια του πουλ των στοιχείων ενεργητικού, εδώ δεν είμαστε υπέρ να, του να είμαστε υπερβολικά παρεμβατικοί. Γιατί αν είναι πάρα πολύ αυστηρός ο κανονισμός, δεν θα αφήσει περιθώρια στα κράτη-μέλη να ορίσουν και αυτά σε ποιο βαθμό θέλουν αυτή την ομογενειοποίηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο για τις μεμονωμένες κατηγορίες των στοιχείων ενεργητικού στο πουλ των ε, στοιχείων ενεργητικού, αλλά θα πρέπει παράλληλα να αφήνουμε στα κράτη-μέλη και τη δυνατότητα να ορίσουν με ποιο τρόπο αυτή η ομοιογένεια θα επιτευχθεί. Θέλουμε δηλαδή να αφήσουμε και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη στο συγκεκριμένο σημείο να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση Επίσης, θέλουμε για τα παράγωγα να τοποθετήσουμε στην οδηγία ένα άρθρο επιπλέον, γιατί πιστεύουμε πως τα παράγωγα επιτρέπουν ε, τα προβλήματα ε, της αναδυστυχίας της νομισματικής μέσα στα στοιχεία ενεργητικού. Και πιστεύουμε πως με μια τέτοια ε, διάταξη ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τα παράγωγα για να σταθεροποιήσουν το πουλ του ενεργετικού. Για την παράταση της οριμότητας, εδώ πάλι έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, γιατί δίνει ε, μία υψηλότερη στάθμιση κινδύνου στις ομολογίες μακρύτερης διάρκειας. Και έχουμε μία σειρά από έγγραφα που αξιοσέβαστα ιδρύματα, στο οποίο λένε πως αυτή η παράταση των ομολογιών ουσιαστικά μειώνει τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, η Moody, η εταιρεία Moody έχει ε, δημοσιεύσει σχετικά άρθρα. Εδώ θέλουμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Λούκη και ίσως εδώ καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ένα κατά αποκοπή συντελεστή που θα σταθμίζει ε, τον κίνδυνο για τα στοιχεία ενεργητικού του πουλ ανεξάρτητα από τη διάρκεια ορίμανσης αυτών. Νομίζω ξεπέρασα το χρόνο μου, οπότε θα σταματήσω εδώ. Thank you very much, Darius. This is my first meeting as, as Vice President. Είναι η πρώτη μου συνεδρίαση σαν uh, αντιπρόεδρος προσπαθήσω λοιπόν να τηρήσω κάποιους κανόνες για το χρόνο. Ο κύριος Αλφρετσάν για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα και βεβαίως ο σκοπός μας είναι να ολοκληρωθεί το θέμα πριν το τέλος της θητείας. Είναι περίπλακο το θέμα και ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αναβολή τελικά. Θα ήθελα εγώ να υποβάλω τροπολογίες, θα σας πω για ποια σημεία, προηγουμένως όμως θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όπως είπατε πρόκειται για εργαλεία, το οποίο ουσιαστικά έχουν βελτιώσει πάρα πολύ σημαντικά την κατάσταση της ρευτότητας και τις οικονομίες της ευρωπαϊκές ε, αγορές καλύπτοντας ε, με ένα σχετικά διαφανές ε, πλαίσιο τους επενδυτές. Οι διασυνοριακές ε, επενδύσεις επίσης έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα στην Γερμανία, τη Δανία. Σήμερα θεωρούνται αυτά τα καλυμμένα ολόλογα πολύ σημαντικά εργαλεία επενδυτικά. Το θέμα λοιπόν που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να μην υπάρχουν υπερβολικές λεπτομέρειες, να δίνεται μία ευελιξία. Η δική μου προσέγγιση όσον αφορά το κείμενο της Επιτροπής είναι το εξής. Αναγνωρίζουμε τις εθνικές πρακτικές και τις διασφαλίζουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο έξυπνοι από τις αγορές. Αυτά λοιπόν που ήδη λειτουργούν και πετυχαίνουν θα τα αφήσουμε να λειτουργήσουν και θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις αδυναμίες και τα ασφάλματα. Όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε στις λεπτομέρειες και να αναθεωρήσουμε αυτά τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί στην Ολομέλεια και να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Ήδη έχουμε υποβάλει σαν Κοινοβούλιο κάποιες ε, τροπολογίες και το θέμα τον ESN πιστεύω ότι πρέπει να μείνει κατά μέρος σε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Θέλουμε φυσικά να προχωρήσουμε βάσει του κειμένου όπως το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Ακούσαμε και τις παρατηρήσεις του εισηγητή όσον αφορά το άρθρο 6 και τα επιλεγμένα στοιχεία του ενεργητικού, το θέμα της ορίμανσης, uh, maturity, και της ε, κατεξουδότηση πράξης. Νομίζω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε κάποια σημεία υπάρχει μεγάλη συμφωνία, ομοφωνία θα έλεγα, για τα παράγωγα και για τις ε, διαρθρωμένες καλυμμένες ομολογίες. Τα θέματα των πουλ, καλυμμένων ομολόγων, εδώ υπάρχει ήδη ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά που ήδη έχουμε ψηφίσει. Στα κοινά καλυμμένα ομόλογα, όπως λέει και ο εισηγητής, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία εγγυώνται τα ομόλογα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι ο κλάδος θέλει να παραμείνει το θέμα των καλυμμένων ομολόγων σαν ένα ξεχωριστό προϊόν και ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ESNs. Εγώ προσωπικά θα έπαιρνα, αν θέλετε, τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού με σκοπό να μην μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες και περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα που αφορά αυτά τα καλυμμένα ομόλογα. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε περισσότερη διαφάνεια στις αγορές και να καλύψουμε και τις ευρωπαϊκές premium καλυμμένες ομολογίες αλλά και τις ε, κρατικές καλυμμένες ομολογίες. Οι προτάσεις μου θα περιοριστούν σε αυτές τις τροπολογίες και δεν θέλω να μπω σε συζήτηση άλλων σημείων για την τροπολογία 13 που δίνουμε ειδική προτιμησιακή αν θέλετε ε, αντιμετώπιση στα λεγόμενα κοινά καλυμμένα ομόλογα αυτά δηλαδή τα οποία δεν έχουν ε, παραπάνω κάλυψη και εγγύησης. Αντίθετα, θα ήθελα εδώ να επανέλθουμε στο θέμα των ε, προθεσμιών της ε, ορίμανσης, maturity, και όσον αφορά τα ποσοστά που ανέφερε ο εισηγητής, θα συμφωνήσω μαζί του για τον κίνδυνο και για την προτιμησιακή μεταχείριση των καλυμμένων ομολογίων. Θα ήθελα να ξέρω από πού προήλθαν αυτά τα ποσοστά σε γενικέ γραμμές το κείμενο της Επιτροπής είναι ένα καλό κείμενο, αν και κάποια σημεία θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε και να τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω και τα σχόλια άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Κάρεναν για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ τον Μπέρναν Λούκε για την έκθεσή του. Υποστηρίζουμε για την πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο τη Καλυμμένη Ομολογία. Σαν τμήμα τη προτάσεω διευρύνεται η ευρωπαϊκή αγορά με τις προτάσεις με σταθερή χρηματοδότηση κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες αγορές. Τα προτινόμενα πλαίσια παρέχουν σε επενδυτές ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον και ευκαιρίε. Αυτό θα προωθήσει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Υποστηρίζουμε τη φύση της προτάσεως. Οδηγία δηλαδή. Έτσι οι εθνικές ιδιαιτερότητες λαμβάνονται υπόψη και ελάχιστη εναρμόνιση ε, πρέπει να γίνει σεβαστή. Όμως, κάποια θέματα υπάρχουν, θεματάκια. Θέλουμε να τα θέσουμε. Εστιαζόμαστε βασικά να είναι ξεκάθαρος ορισμός των καλυμμένων ομολόγων. Αυτό σχετίζεται με το άρθρο 6 και τα ανέφερα αυτό και συνάδελφοι. Το άρθρο 6 έχει πολύ χαμηλά όρια. Πρέπει να αναφέρονται τα ποιοτικά αξιόγραφα που ξεπερνούν τα όρια του CRR. Πρέπει να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές τα καλυμμένα ομόλογα. Να αποφύγουμε από δυνάμωση της ποιότητας των καλυμμένων ομολόγων, της κατηγορίας αυτής των αξιογράφων. Αναγνωρίζω ότι αυτό ξεπερνά τις τροπολογίες που υπέβαλε ο εισηγητής Εκτιμώ όμως την προσπάθεια που κατέβαλε να διαφυλάξει την ποιότητα ε, της ε, κατηγορίας αυτής των καλυμμένων ομολόγων. Τροπολογίες δεν υποστηρίζω κάποιες ομολογίες, όπως οι 4 και 5 του κανονισμού. Αυτές οι τροπολογίες θέλουν να θεσπίσουν υψηλότερη στάθμιση κινδύνου για κάποια καλυμμένα ομολόγα, με επεκτάσιμες οριμότητες. Οι προτάσεις βαθμολόγησης με τριπλό αλφα για τα καλυμμένα ομόλογα CPT είναι σε μειονεκτική θέση. Έναντι χαμηλότερων ή ποιοτέρων ε, ομολόγων τύπου soft bullet. Η στάθμιση του κινδύνου για βαθμολόγηση 3α CPT ομολόγων καλυμμένων θα πήγαινε από 10% στο 13%. Και αυτή η πρόταση διαταράσσει μια εύρυθμα αγορά και αυτό δεν στηρίζεται από τα στοιχεία που έχουμε από την αγορά. Υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για τα καλυμμένα ομόλογα. Για να διατηρηθεί η ποιότητα αυτής κατηγορίας αξιογράφων και θέλουμε να επιτρέψουμε να ληφθούν υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες. Προσβλέπω στις μελλοντικές συζητήσεις των σκιωδών και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το, της εργασίας επί του θέματος πριν από το τέλος της αιτίας και κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Καρολάιν. Ο Φιλίπ Λαμπέρ, εκ μέρους των Πρασίνων, ζητάει συγγνώμη που δεν θα μιλήσει. Μετά Γκουε. Μαρίσα, Ματέος. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλιστή. Ah, eu, vou fazer um comentário muito global em relação às propostas que estamos a discutir. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση γενικότερη για τις προτάσεις αυτές συζητάμε και ελπίζω πως ε, ο συνάδελφος εισηγητής θα βάλει τα ακουστικά για να με ακούσει. Να σας πω το εξή. Αργότερα εγώ θα καταθέσω τροπολογίες πολύ πιο συγκεκριμένες, αλλά έχω μια γενική παρατήρηση για τα όσα έχω να σας πω ε, για το κείμενο και συμφωνώ με τον εισηγητή, με τον Μπέρντ Λούκε, γιατί στην αιτιολογική έκθεση μιλά για ομολογίες εγγυημένες και καλυμμένες και τις χαρακτηρίζει αντίθετα με άλλα είδους εργαλεία ως εργαλεία στέρεα που μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ο κανονισμός σχετικός με αυτά τα ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία να μην υποπέσει στο εξή φάλμα, Να ρυθμίσει κάτι και να φτιάξει κάτι το οποίο δεν είναι χαλασμένο. Δηλαδή πιστεύω ότι πως αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να προωθηθούν, θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθεί ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ίσως να περιμένουμε και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε λίγο αυτά τα οποία παρουσιάζει ο εισηγητής. Ε, θα καταθέσω τις σχετικές τροπολογίες αργότερα, αλλά έχω κάποιες ανησυχίες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Καταρχήν, τα κανονιστικά ή ρυθμιστικά προβλήματα από το γεγονός πως έχουμε ενστοιχεία ενεργητικού που συμπεριλάβουμε που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της διασύνδεσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών συστημάτων υπάρχει ακόμα το θέμα που είναι ε, τι συμβαίνει με, αυτά τα, με αυτές τις ομολογίες και τις καλυμμένες ομολογίες, οι οποίες όμως ρυθμίζονται από πλαίσια ε, ρυθμιστικά ε, που δεν είναι ε, ενουσιακά. Από αυτό περνάω στο επόμενο σημείο που είναι τα παράγωγα και το πώς θα καλύψουμε εκεί τους κινδύνους και αν θα χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ πως είναι κάπως αφελές να θεωρούμε πως αυτός είναι ο τρόπος για να καταφέρουμε αυτό το οποίο επιδιώκει το έγγραφο μπροστά μας. Γιατί αν δείτε τι συζητήσεις έγιναν από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, και επαναλαμβάνω, θα τα πω πιο συγκεκριμένα στι τροπολογίε μα. Πιστεύω λοιπόν πω το να συμπεριλάβουμε τα παράγωγα σε αυτά τα καλυμμένα στοιχεία ενεργητικά απλώ είναι ένα υποκατάστατο το οποίο δεν γίνεται την κατάλληλη στιγμή Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει μια πραγματική αξιολόγηση κινδύνου και να μα δώσει την πραγματική ασφάλεια και σταθερότητα παρά μόνο δημιουργεί μια πλασματική ασφάλεια ε, η οποία εμένα με ανησυχεί και είναι από τα κεφάλαια στα οποία θα υποβάλω τι πιο πολλέ τροπολογίε. Ξέρω πω είναι διαφορετικέ οι θέσει σα, αλλά επαναλαμβάνω, είμαι ε, πραγματικά στη διάθεσή σα για να συνεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε κάποια μέτρα και κάποιε συναλλαγέ ε, που ε, θα καλύψουν και τι δικέ μου ανησυχίε και τι ανησυχίε των υπόλοιπων σχεδόν εισηγητών. Δυστυχώ θα χρειαστεί να φύγω από την αίθουσα, γιατί πρέπει να πάω και στην Επιτροπή Ήτρε, γιατί έχουμε το Horizon 2020, ε, οπότε ε, γραπτά τα υπόλοιπα σχόλια. Uh, Ευχαριστώ πολύ Μαρίσα. ΕΝΕΦ. Η Μπάρμπαρα Κάπελ είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Ωραία. Πάμε στη δικασία Καστιάη. Ένας έχει ζητήσει το λόγο. Ο συντονιστής των συλλιστών, υπερβόνς, υπερβόνς Περές, έχει το λόγο. Euh, Συγχαρητήρια, Πρόεδρε, για την ε, πρώτη άσκηση αυτή, η πρώτη ημέρα άσκησης των καθηκόντων σας. Και που κατευθύνει τι συζητήσεις μας. Πολλά υπόθηκαν. Και οι σκιώδεις ηγητές πολλών ομάδων εξέθεσαν το θέμα. Και κάλυφθηκαν οι ανησυχίε μου. Επιμένω επί του πνεύματος επί του που εργαστήκαμε όσον αφορά την έκθεση πρωτοβουλία. Βρήκαμε έναν τρόπο να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που δίνει προστιθέμενη αξία, χωρί να καταστρέφουμε αυτό που λειτουργούσε. Κυρίω τα εθνικά καθεστώτα. Όταν επιτρέπω μια χρηματοδότηση μέσω αυτού του εργαλείου, του covered bond, μηχανισμού που είναι αποτελεσματικό. Είχαμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν επακριβώ όπως έκανε και ο κύριος Σάντζος και ο δισηγητής και ο Ντάριος Ροζάτη τα είπαν αυτά. Τώρα, όσον αφορά τις συστάσεις που με υπόψη για το μεικτό χαρακτήρα κάποιων covered bond υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούν στις διάφορες αγορές και θα πρέπει να συνεχιστούν. Και το θέμα της ε, αντιατάραξης του χαρακτηριστικού της οριμότητας. Αυτά που είπε ο Ντάριους Ροζάτη ήταν σωστά. Αυτά είναι κάποια σχόλια που είχα. Ο εισηγητής θα θέλει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Πρέπει να διευρυνθεί όμως η βάση διαπραγματεύσεων για να συμπεριληφθούν οι διάφορες ε, ιδέες οι οποίες είχαν αναφερθεί στην έκθεση ιδέε πρωτοβουλία συμπεριληφθούν και εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Περβάνς. Ε, άλλος συνάδελφο που θέλει να μιλήσει. Δεν υπάρχει άλλος που θέλει να χορεύσει. Κύριε Λουκ, μπορείτε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ τους για τα σχόλια που κάνατε στην έκθεσή μου. Χαίρομαι για τις ε, γενικές γραμμές. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω, η ιδέα της διάκρισης μεταξύ των ε, premium και των κοινών ε, καλυμμένων ομολόγων είναι κάτι που τουλάχιστον βρίσκει σύμφωνους όλους όσους πήραν το λόγο. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συνένεση και στο θέμα της ε, ειδική ε, μεταχείρισης, προτιμησιακής μεταχείρισης των ε, κοινών καλυμμένων ομολόγων και αυτό το θεωρώ ένα είδος καλής προϋπόθεσης για να ξεκινήσουμε. Επίσης το θέμα των ESN, λυπάμαι που πρέπει να τα εγκαταλείψουμε, αλλά πιέζει ο χρόνος και βλέπω ότι συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο, όπως παραδείγματος χάρη το άρθρο 6, 6α στην έκθεσή μου, που θέτει πολύ χαμηλά το όριο, όπως είπε η Κάρολάιν. Επίσης, ακούσαμε και τα καλυμμένα ομόλογα και τις ε, προϋποθέσεις της 129 όπως ε, είπατε εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας αρχικά δεν θέλαμε να είμαστε πολύ επεμβατική στην αγορά. Και ουσιαστικά εδώ παίρνουμε και ασχολούμαστε μόνο με ένα υποσύνολο των ε, καλυμμένων ομολόγων. Υπάρχουν και κάποια άλλα καλυμμένα ομόλογα που θα πρέπει να τηρούν λιγότερες από τις 129 προποθέσεις. Ουσιαστικά εδώ το άρθρο 6α δίνει μια πιο συγκεκριμένη έννοια αυτό του πουλ των καλυμμένων ομολόγων που δεν αναφέρονται ρητά στην άλλη διάταξη. Αυτό το άρθρο λοιπόν 6α ε, και αν το όριο τίθεται πολύ χαμηλά, άκουσα την ΚΟΕ. Η ΚΟΕ θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλά το όριο ε, στο 6. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό γιατί σαφώς ε, φαίνεται εδώ ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Εγώ ήθελα όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτουν αυτά τα ομόλογα ήθελα να θέσουμε κάποια ποιοτικά κριτήρια πολύ συγκεκριμένα. Ίσως όμως χρειάζεται περισσότερη συζήτηση μεταξύ των σκιωδών ε, εισηγητών για το άρθρο 6α. Θα δούμε. Κάποιες ε, προτάσεις που κάνω για κάποια στάθμιση κινδύνου, ιδιαίτερα για την παράταση της ε, ημερομηνίας ορίμανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει τέτοιου είδους προτάσεις για το θέμα αυτό. Εγώ θα μπορούσα ενδεχομένως να είχα υποβάλει τροπολογίες μην χωρίς να είμαι συγκεκριμένος στους αριθμούς βάζοντας χιχιχι ή κάτι άλλο στη θέση των αριθμών. Ήθελα παρόλα αυτά να υποβάλω κάποιες ρεαλιστικές σταθμισμένες προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο υπάρχον πλαίσιο ρυθμιστικών κανόνων, αυτών δηλαδή που υπάρχουν και ισχύουν, χωρίς να δημιουργήσω την οποιαδήποτε ε, διαταραχή. Επίσης ε, υπάρχουν σήμερα κάποια ποσοστά, το 80%, το 60% που ο Δάριος Τροζάτη ανέφερε. Πρόκειται για, θα έλεγα, μετριοπαθείς προτάσεις, προτάσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τα στοιχεία, τα περιουσιακά, πώς ενσωματώνονται και ποια είναι τα ποσοστά για την στάθμιση κινδύνου επαναλαμβάνω, στο CRR υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού τα οποία λαμβάνονταν υπόψη. Εγώ ήθελα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να δείξω ότι αυτές οι προτάσεις που επαναλαμβάνω είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, οι συζητήσεις με τους κοιόδες θα συνεχιστούν, ο τριμερής διάλογος ε, θα αποτελέσει μια αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση. Πρόκειται για αριθμούς, πρόκειται για ποσοστά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τελική αυτή η αριθμή. Θα τους ξανασυζητήσουμε με τους κοιόδες ηγητές. Τώρα, αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να περιπλέξουμε περισσότερο το σύστημα, δεν πρέπει να μπούμε σε υπερβολικές ε, λεπτομέρειες. Οι αγορές λειτουργούν, μια χαρά λειτουργούν. Δεν πρέπει λοιπόν να τις διαταράξουμε. Κάποιες από τις νέες ιδέες που περιέχει αυτή η έκθεση έχουν προέλθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως προσθέτουν κάτι στον κανονισμό μας. Δεν υπάρχουν στον κανονισμό μας δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία, τα οποία τα έχει υποβάλει η Επιτροπή, εντελώς νέα στοιχεία. Εγώ μπορώ να σβήσω κάποιες από αυτές τις ιδέες, όπως παραδείγματο χάρη η ιδέα της κοινή χρηματοδότησης. Αν δεν συμφωνούσε μπορούμε να το διαγράψουμε. Κοινή χρηματοδότηση, κοινή διασυνοριακή χρηματοδότηση. Αυτό πιστεύω εγώ ότι εάν παραμείνει στην έκθεση πρέπει να διευκρινιστεί πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει η Επιτροπή. Τώρα για τα παράγωγα. Εδώ μπορούμε ενδεχομένως να συζητήσουμε τη διατύπωση πιο πολύ, όχι τις έννοιες. Σίγουρα η στάθμιση του κινδύνου, η οποία γίνεται μέσω αυτών των παραγόγων προϊόντων, μέσω των εγγυήσεων, και ακριβώς η έκδοση αυτών των καλυμμένων ε, ομολόγων, τα παράγωγα όπως διατυπώνονται εδώ, γι' αυτό και επαναλαμβάνω, είναι θέμα διατύπωσης πιο πολύ παρά ενιών. Το αν δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού αυτού μπορεί να διατυπώνονται και να εκφράζονται σε συναλλαγματικές ε, ισοτιμίες σε διαφορετικά νομίσματα κτλ. κτλ. Επαναλαμβάνω εδώ χρειάζεται διευκρίνηση και καλύτερη διατύπωση. Ο Τάριος Ροζάτη επίσης αναφέρθηκε στις εγγύησει σε ποιο είδος στάθμισης κινδύνου θέλουμε να φτάσουμε, αν υπάρχει το λεγόμενο flat risk, και αν υπάρχουν προθεσμίες, δηλαδή για την πρώτη διετία και για την επόμενη περίοδο. Εγώ ενδεχομένω θα δεχόμουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σχόλια. Α, η ομοιογένεια. Δεν μίλησα για την ομοιογένεια. Και αυτό είναι η ιδέα της Επιτροπής. Εγώ αυτή την προϋπόθεση δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να τη δεχτώ γιατί η ομοιογένεια από τη μία μπορεί να βοηθάει ενδεχομένως την ανάλυση των επενδυτών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Από την άλλη, η ετερογένεια είναι εξίσου ελκυστική. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πλήρης ομοιομορφία στην αγορά. Δεν νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πλήρη ομοιογένεια και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θέλουμε να προχωρήσουμε και να ακολουθήσουμε αυτή την ε, πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούκε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε και το χρονοδιάγραμμα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Βεβαίως ακούσαμε κάποιες παρουσιάσεις φέτος. Και να σας πω πως η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 Σεπτεμβρίου στις 5. Θα τις συζητήσουμε στις 18 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 25 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, η προηγούμενη ημερομηνία λοιπόν ήταν του Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε 5 Νοεμβρίου. 18 λοιπόν Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε, 18 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο 6, διάφορα, δεν βλέπω κάτι. Άρα λοιπόν η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στις 3 στις Βρυξέλλες. Γεια σας.